Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι δήλωση Αντιπροέδρου της Επιτροπή, υπάτηση εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Θέμα η κατάσταση στην Συρία. Ο κύριος Ανδρέας Μαυρογιάννης, εκπρόσωπος της Προεδρίας, έχει το λόγο εξ ονόματος της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και υπάτης εκπροσώπου. Κύριε Υπουργέ. Κύριε Πρόεδρε, έντιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με μεγάλη χαρά σας παρουσιάζω τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις πρόσφατες δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Συρία εξ ονόματος της ΥΠΑ του εκπροσώπου και αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Κάθριν Άστον. Η κατάσταση στη Συρία εξακολουθεί να δίνει λαβή για συνεχιζόμενες ανησυχίε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η βία έχει οξυνθεί, ο αριθμός των θυμάτων έχει φτάσει απίστευτα ύψη. Ο κίνδυνος ενό εμφυλίου πολέμου έχει γίνει πιο απτός και πραγματικό, και υπάρχουν ήδη ενδείξεις για συγκρούσεις μεταξύ ομολογιακών ομάδων και πολιτικών αντιμετώπων ομάδων. Μια επέκταση αυτή τη σύραξη θα έχει σημαντικέ επιπτώσει όχι μόνο για τη Συρία αλλά και για τη σύνολη περιοχή. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ενισχύσει τι δραστηριότητε για τη Συρία με στόχο να μπορέσουν το ταχύτερο δυνατόν να σταματήσουν οι εχθροπραξίε και η βία και να βρεθεί μια λύση η οποία θα οδηγήσει σε μια ειρηνική πολιτική μετάβαση στη Συρία με την πρωτοβουλία των ίδιων των Σύριων. Η τρέχουσα εβδομάδα είναι ιδιαίτερα έντονη γιατί συνεχίζονται οι προσπάθειες σε διεθνές επίπεδο για να υπάρξει μία ενίσχυση και εδραίωση και ενοποίηση της διεθνούς απάντησης στα προβλήματα της κρίσης στη Συρία. Αυτά ακριβώς τα ανέφερε και η κυρία Άστον εδώ στην, προσ... στην προηγούμενη Ολομέλεια ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρξει ένα οδικό χάρτη ο οποίο θα υποστηρίξει τον Κόφι Ανάν, θα ενισχύσει τη διεθνή παρουσία και θα κάνει πιο ενιαίε και πιο ανθεκτικέ τι διπλωματικέ προσπάθειε, κάτι το οποίο συμπεριλαμβάνει και την έκκληση για δράση του Συμβουλίου Ασφαλεία και τη συμμετοχή τη Ρωσία και τη Κίνα. Η υπερδιεκπρόσωπο και αντιπρόεδρο Κάθη Άστον ήταν παρούσα στην συνεδρία τη Γενέβη για την ομάδα δράση για τη Συρία που είχε ε, συγκληθεί από τον ειδικό από απεσταλμένο του ΟΗΕ τον Κόφι το προηγούμενο Σάββατο. Όπως γνωρίζετε, με παρουσία του ΟΗΕ, του Αραβικού Συνδέσμου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κίνας, της ε, Ρωσίας, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, Ηνωμένων Πολιτειών, Τουρκία, Ιράκ, Κουβέιτ, συμφώνησαν σε βασικές αρχές και κατευθυντήριε γραμμές για μια μετάβαση με ηγεσία των ίδιων των Συρίων που θα οδηγούσε στη δημιουργία ενός μεταβατικού κοινοβουλευτικού σώματος το οποίο θα είχε πλήρε εξο... εκτελεστικές εξουσίες. Μια μάλλον κοινοβουλευτική αλλά κυβερνητική, ε, κυβερνητικό φορέα. Θα μπορούσε λοιπόν με αμοιβαία συμφωνία να δημιουργηθεί αυτή η κυβέρνηση. Η ομάδα δράση επίση, υποστήριξε ανέφερε ότι υποστηρίζει πλήρω τον Κόφι Ανάν και το έξι σημείων σχέδιό του. Σε ό,τι αφορά την αποστολή παρατήρησης των Ηνωμένων Εθνών στην Συρία, έχει πάρει νέα ορμή και όθηση χάρη στις προσπάθειες του ειδικού απεσταλμένου. Επίσης, ε, είναι προσιλωμένες και δεσμευμένες οι δυνάμεις αυτές, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ο Αραβικός Σύνδεσμος της Ευρώπη κτλ. στο να αντισταθούν σε οποιαδήποτε κλιμάκωση της βίας. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν εφαρμογή αυτών των μέτρων, γιατί όλα αυτά είναι θετικά μέτρα και πρέπει συνολικά και συλλογικά να εξασφαλίσουμε ότι θα υλοποιηθούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δεσμευμένη να πράξει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να προωθηθεί αυτή η διαδικασία. Στην συνέχεια, μετά από την ομάδα ε, ε, Επαφή στην Γενέβη θα συναντηθούν οι φίλοι της Συρίας στο Παρίσι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι παρούσα σε αυτή τη συνάντηση όπου θα συμμετέχουν μέχρι και 100 χώρες. Η ελπίδα μας είναι ότι η συνάντηση των φίλων της Συρίας θα επικυρώσει την προσπάθεια της ομάδας δράσης για να υπάρξει μια κοινή απάντηση από τη διεθνή κοινότητα. Έχουμε μεγάλες προκλήσεις για να εφαρμοστούν αυτές οι αρχές σε μια πραγματική μεταβατική διαδικασία. Υπάρχουν κέρια θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν όπως είναι η ανάγκη να υπάρξει και ένας εντεταλμένος <clears throat> συνομιλητής από την Συριακή κυβέρνηση ο οποίος να είναι αποδεκτός και στην αντιπολίτευση. Πολλές πτέρυγες αντιπολίτευσης δεν είναι έτοιμες ούτε καν να διαπραγματευτούν, επομένως είναι δύσκολο να επιτύχουμε μια πολιτική λύση. Η αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των βημάτων απαιτεί επίσης μια συνεκτική και αντιπροσωπευτική αντιπολίτευση. Η συνάντηση που έγινε στο Κάιρο, οργανωμένη από τον Αραβικό Σύνδεσμο των Ομάδων της Αντιπολίτευσης και με παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν ένα ακόμα θετικό βήμα για να προσπαθήσουμε να συνενώσουμε τις διάφορες αντιπολιτευτικές ομάδες. Πρέπει να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ των απόψεων των διαφορετικών ομάδων αντιπολίτευσης μέσα στη Συρία και αυτών που βρισκόνται εκτός Συρίας. Πρωτοβουλία <clears throat> τη ΥΠΑ του εκπροσώπου και αντιπρόεδρου κυρία Άστον, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να συναντάται με εκπροσώπους διαφόρων ομάδων στη Συρία έχουν υποστηρίξει και έχουν χρηματοδοτήσει σεμινάρια στις Βρυξέλλες από το μέσο σταθεροποίησης που οργανώνονται υπέρ των Συρίων για τα θέματα μετάβασης. Το πρώτο σεμινάριο που έλαβε χώρα στις 24 25 Ιουνίου στις Βρυξέλλες συνένωσε μια μεγάλη πλειάδα προσωπικότητων τη αντιπολίτευση για να συζητήσουν θέματα που έχουν να κάνουν με τη διαδικασία μετάβαση και αυτό περιλαμβάνει στις συνταγματικές και υπερεθνικές αρχέ, οικονομικέ και αρχέ και κοινωνικέ αντιμετωπίσει και φυσικά τα δικαιώματα των μειονοτήτων στη Συρία. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά όπως έχει επιστήσει την προσοχή μας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανειλημμένα. Το μήνυμα λοιπόν της ΥΠΑ του εκπροσώπου είναι ότι η Συρία είναι για όλους τους Σύριους συμπεριλαμβάνοντα και όλε τι μειοψηφίε των οποίων τα δικαιώματα θα πρέπει να τύχουν σεβασμό. Το δεύτερο σεμινάριο αυτού του είδου θα γίνει στα μέσα Ιουλίου στο Κάιρο. Η, τα σεμινάρια αυτά για τους εκπροσώπους τη αντιπολίτευσης συμβάλλουν σε μια πολιτική διαργασία η οποία έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει τη διαμόρφωση μιας αντιπροσωπευτικής αντιπολίτευσης. Με τον τρόπο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει ρόλο διευκολυντή για να υπάρξει ένα περιεκτικός διάλογο που να έχει ηγεσία από τους ίδιους τους Σύριους και η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να ζητά να υπάρχει ενιαία δράση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Εθνών για να μπορέσει να ασκηθεί αποτελεσματική πίεση στο καθεστώς της Συρίας. Είναι μεγάλη η ευθύνη της κυβέρνησης της Συρίας για τη βία η οποία έχει ασκηθεί, συνεχίζονται οι σφαγές ενώ οι διεθνείς προσπάθειες είναι ακόμα εν εξελίξη. Όλα αυτά είναι απαράδεκτα και αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για αυτά τα εγκλήματα στην τωρινή αυτή αντιπαράθεση θα πρέπει να λογοδοτήσουν γι' αυτό. Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν περιορίζεται στη διπλωματία και την πολιτική διαδικασία σε όλα τα επίπεδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να αυξάνει τις ενέργειές της και να ασκεί κυρώσεις όσο συνεχίζει αυτή η κατάσταση. Οι κυρώσεις αυτές στοχεύουν στην κυβέρνηση της Συρίας για να μπορέσουν να μειώσουν τους πόρους τους αλλά με ελάχιστη επίπτωση στον πληθυσμό της Συρίας. Πρόσφατα αποφασίστηκε ένας νέος γύρος κυρώσεων που έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία από το Μάιο του 2011. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τώρα να ε, συνεννοούμεθα με τους εταίρους μας για να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των κυρώσεων και να συνεχίσουμε τη διεθνή πίεση κατά της Συρίας. Η διμέρης βοήθεια βέβαια έχει ανασταλεί, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει υποστήριξη σε μία πλειάδα <clears throat> οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στις 8 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε ένα πακέτο υποστήριξης 23 εκατομμυρίων ευρώ για να υποστηρίξουν και την κοινωνία των πολιτών στη Συρία και τους πρόσφυγες στις όμορες χώρες σε περιοχές οι οποίες έχουν επηρεαστεί από την εισρωή προσφύγων από τη Συρία. Η ανθρωπιστική πρόσβαση παραμένει ένα θέμα ανησυχίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να παρακολουθεί την εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της Συριακής Κυβέρνησης και, και του ΟΗΕ πολύ προσεκτικά. Μέχρι στιγμής η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει πάνω από 44,6 εκατομμύρια ευρώ για να αντιμετωπιστούν ανθρωπιστικές ανάγκες μέσα στη Συρία και στις όμορες χώρες. Εν τέλει, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει την ε, αποστολή παρακολούθησης του ΟΗΕ με 8,2 εκατομμύρια ευρώ. Τα κονδύλια αυτά χρηματοδοτούν 25 θωρακισμένα οχήματα, την επιμελητία και την υποστήριξη για δυνατότητα χρήσης ασθενοφόρων αν αυτό απαιτηθεί. Και υποστηρίζει μια περιεκτική διαδικασία διαλόγου που μπορεί να βοηθήσει την επίτευξη πολιτικής λύσης στη Συρία. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω έντιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει τις προσπάθειές της και δεν θα αφιστεί προσπαθειών για να υποστηρίξει τον λαό της Συρίας στον αγώνα του για ελευθερία και ειρήνη και για να διευκολύνουμε μια ειρηνική μετάβαση στη χώρα αυτή. Ευχαριστώ πολύ. ευχαριστούμε κύριε Μακρογιάννη. Ακολουθούν τώρα οι ομιλητέ εξ ονόμων των ομάδων. Η κυρία Ντεκάιζερ. Πόσο χρόνο έχω? Δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως υποστηρίζουμε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασκείται από την κυρία Άστον. Όμως, σήμερα ψάχνω μέσα στα μετριοπαθή μέσα που έχουμε στα, μέτρια μέσα που στη διάθεσή μας, τι είναι διαθέσιμο, τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διότι συζητούνται στους διάφορους κύκλους, στους ύψιστους κύκλους ε, το τι μπορούμε να κάνουμε, εμείς τι μπορούμε να κάνουμε. Και εδώ και τρει εβδομάδες ε, τον Λαμποάνη, έναν ιστορικό αντιπολιτευόμενο της Συρίας που είχε φυλακιστεί εδώ και πέντε χρόνια, όταν εγκατέλειψε από το κοινοβούλιο, πήγε στη Δαμασκό και φυλακίστηκε αμέσως. Δεν ήταν και ο πρώτος που φυλακίστηκε. Και στο γραφείο μου εδώ και πέντε χρόνια συζητούσαμε μαζί τις συνθήκες που επικρατούσαν στις φυλακές της, ε, του Μπασάρα Ρασάντ και μιλούσαμε για τις απόπειρες αυτοκτονίας. Ε, είπε ήταν φρικτά, του είπα δεν φοβάται, είπε όχι δεν θα αυτοκτονούσα. Με συγκίνησε όταν επανήλθε και μου είπε κυρία Ντεκάιζερ ε, δίδατε δεν αυτοκτόνησα και σήμερα ζω το πιο το πιο ωραίο κομμάτι τη ζωή μου που δεν φαντάστηκα ποτέ ότι θα ζούσα. Και ανεξάρτητες φαγές που γίνονται σήμερα, ποτέ δεν είχα φανταστεί ότι θα έβλεπα αυτέ τι μέρε στη Συρία. Άρα πέρα τι φαγές, πέρα από τι από τις φρικαλαιότητες που λαμβάνουν χώρα, υπάρχει ελπίδα στο πληθυσμό των πολιτών σήμερα στην Συρία που δεν πρέπει να απογοητεύσουμε. Και είπα τι μπορούμε να κάνουμε όταν άκουσα αυτό το μήνυμα. Αυτό ε, με διακατέχει. Έχω μπροστά μου την έκθεση του Human Rights Watch και του Amnesty International. Έχω, βλέπω όλα αυτά που καταμετρούνται όσον αφορά τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, τα βασανιστήρια σήμερα που γίνονται στη Συρία και δεν τολμώ καν, Πρόεδρε, να σας διαβάσω αυτές τις μαρτυρίες γιατί ε, ξεπερνά την έκπληξη θέλω να σας πω ότι πρέπει να ετοιμάσουμε αυτό που θα ακολουθήσει τον Μπασάρ Ρασάτ Θα πρέπει ε, να ακούσουμε τις μαρτυρίες, να επιχειρηματολογήσουμε. Το ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διακόπτω το μικρόφωνο τη ομιλήτριας. Ευχαριστώ. Ακολουθεί κυρία Σάκε για δύο λεπτά. Όχι, όχι, όχι. όχι, όχι. Λυπάμαι κυρία Δεκέιζερ Είχατε δύο λεπτά και αρχίσαμε το ρολόι όταν αρχίσατε να μιλάτε. Λυπάμαι, κυρία Σάκη. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Πέρασαν έξι εβδομάδες από όταν είδαν σφιχτές εικόνες από τα σφαγή στη Χούλα. Είδαμε δολοφονημένα παιδιά και θεωρήσαν ότι ήταν και το σημείο μια επιστροφή Τότε είδα κάποιοι. Και, είπαν... και ακούστηκαν τα λόγια ποτέ ξανά. Συνεχίζει τον πόλεμο το καθεστώς Ασάντ κατά του πληθυσμού της Συρίας και πολλοί όμως γενναίοι Σύριοι είναι πρόθυμοι να πληρώσουν το ύψιστο τίμημα όταν διαμαρτύρονται ειρηνικά για την ελευθερία και το σεβασμό της αξιοπρέπειάς τους και των δικαιωμάτων τους. Ε, διάφοροι στατιωτικοί ε, που ε, ξέφυγαν είπαν ότι βασανίστηκαν, διάφοροι διάλεξαν να αυτοκτονήσουν και θα πρέπει να δείξουμε στο συριακό πληθυσμό ότι δεν του δυσμονήσουμε. Έχουμε ευθύνη να προστατεύσουμε και τι σημαίνει αυτό. Η λύση στη Συρία δεν είναι εύκολος. Η νέα ομάδα δράση για τη Συρία ντόπισε βήματα για την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου του Κόφι Ανάν με τα σημεία και του ψηφίσματο του ΟΗΕ. Οι προσπάθειε αυτέ θα πρέπει να υλοποιηθούν το ταχύτερο δυνατόν. Δεν πρέπει όμω να αφαιρούμεθα το στόχο και καλωσορίζω τη συγκρατημένη ανταπόκριση της Τουρκίας παρά ε, την πρόκληση της Συρίας που κατέριψε το αεροσκάφος στρατιωτικό και που σκοτώθηκαν οι δύο πιλότοι. Και απευθύνω τις σκέψεις μου και απευθύνω προς τις οικογένειες αυτών των πιλότων. Λυπούμε ότι τελικά είδαμε ότι επικρατούν συμφέροντα εντό ζώων των ανθρώπων και πλευρά Ρωσία. Όμω και η Ρωσία θα πρέπει να αποτελέσει κομμάτι τη λύση στην κρίση, όσο και δύσκολο και σκληρό αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίω επί Κυπριακή Προεδρία, ε, πρέπει να δούμε ότι έχουμε τεράστιες ευθύνες και θα πρέπει να κάνουμε ανοιχτές διαφανείς έρευνες για το πώς ένα ρωσικό πλοίο που μετέφερε όπλα μπορεί να φτάσει στις ακτές της Συρίας αφού ε, ελιμενίστηκε σε κυπριακό λιμάνι και αφού εντοπίστηκε από τις κυπριακές αρχές. Αυτό το κοινοβούλιο ζήτησε από δικά να ξεκινήσει πλήρη έρευνα, αλλά μέχρι τώρα δεν έχουμε πραγματικές διαβεβαιώσεις όσον αφορά το γεγονός όταν οι κυρώσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εφαρμόζονται, είναι μόνο άσκηση επιχάρτου και δεν καθησυχάζουν το λαό τη Συρία. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Σάκε, ακολουθεί η κυρία Φλότρο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ η κυρία Σάκε. Αντιμετώπισε ένα θέμα το οποίο είναι πραγματικά ιδιαίτερα εύστοχο και πιστεύω ότι θα απαντήσει για το θέμα αυτό η Προεδρία του Συμβουλίου. Η κατάσταση η επιτόπια κατάσταση όπως έχει παρουσιαστεί έχει φτάσει την κορονίδα της βίας, έχει φτάσει μια αποκαλυπτική βία πια. Είχαμε μόνο την προηγούμενη εβδομάδα 800 νεκρούς. Η έκθεση του Human Rights Watch λέει ότι σε 27 κέντρα κράτησης υπάρχουν συστηματικά βασανιστήρια και οι μαρτυρίες είναι συντριπτικές. Βλέπουμε εδώ και μια εβδομάδα νέες πρωτοβουλίες σε διπλωματικό επίπεδο, οι οποίες ίσως προϊονίζονται στοιχεία μιας αλλαγής στην κατεύθυνση για την επίτευξη μιας λύσης. Πιστεύω ότι η συνάντηση της Γενέβης ήταν μια απαρχή ακόμα και περιορισμένη για να μπορέσει να προκύψει μια μεταβατική κυβέρνηση εθνικής ενότητα στη Συρία χωρίς τον Ασάντ και τους βασανιστές του. Αυτό θα έχει δύο σε αυτή την κατάσταση. Όχι επειδή υπάρχει η προοπτική μιας λύσης θα μειωθεί η βία ίσα ίσα θα υπάρξει μια όξυνση της βίας κατά πιθανότητα από την πλευρά της κυβέρνησης. Αλλά η προοπτική αυτή οδηγεί σε όλο και περισσότερες λιποταξίες των στρατιωτικών από το καθεστώς του Ασάτ και θα επιτρέψει σε αυτό το μεταβατικό ε, σχέδιο να υπάρξουν και κάποιοι οι οποίοι είχαν υποστηρίξει προηγουμένως τον Ασάτ μέσα στο κόμμα Μπαάθ. Είναι λοιπόν πάρα πολύ κέρια αυτή η χρονική στιγμή. Εγώ θα ήθελα αυτή η προοπτική η οποία είχε υποστηριχθεί από την συνάντηση όλων των ε, συνιστοσών της αντιπολίτευσης της, στη Συρίας με τον Αραβικό Σύνδεσμο ότι θα οδηγήσουν σε μια αλλαγή, ότι θα υπάρξει μια τροποποίηση της κατάστασης και θα ανοίξει λοιπόν ένα μικρό παράθυρο ελπίδας για το μέλλον και εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διαδραματίσει πλήρως το ρόλο της όπως θα πρέπει να κάνει και στο Σαββατοκύριακο στο Παρίσι τη συνεδρίαση των φίλων της Συρίας, του λαού της Συρίας συγκεκριμένα. Ευχαριστώ κύριε Φλότρο. Ο κύριος Φαν Όρτεν για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, δυστυχώς γνωρίζουμε τις ακρότητες και το ανθρώπινο κόστος της κατάστασης στην Συρία και το φοβερό αντίκτυπο στο συριακό λαό. Εγώ θέλω να εστιαστώ σε ευρύτερες συνέπειες για την περιφερειακή ασφάλεια. Η Συρία βεβαίως ε, εδώ και καιρό ήταν ε, πάρα πολύ, είχε πάρα πολύ στενές σχέσεις με το καθεστώς του Ιράν, προωθούσε την τρομοκρατία σε άλλες χώρες. Πρόσφατα η Χαμάς πήρε το αρχηγείο της και μετακόμισε από τη Δαμασκό και βεβαίως υποδέχονταν και το ΠΚΚ ο Ασάντ και είχε βεβαίως βάσεις επιμελητίας, είχε Σμπολάχ και άλλες ε, οργανώσεις ε, με τρομοκρατικούς κλάδους. Βεβαίως ε, υπήρχε και πρόβλημα με την ειρήνη με το Ισραήλ καθώς τα σύνορά τους συνεχώς απειλούνταν από συριακές ε, επιθέσεις και από οργανώσεις που στήριζε και βεβαίως θα πρέπει να φροντίσουμε η Συρία να μην αποτελεί μέρος στο οποίο βρίσκουν καταφύγιο τρομοκρατικά κινήματα και πρέπει να βοηθήσουμε τις ε, δύο χώρες για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που έχουν από την βία του Ασάτ. Σας ευχαριστώ κύριε Φαν Όρντεν. Δυστυχώς ο κύριος Αγκουράκης δεν είναι εδώ. Οπότε ο κύριος Σκοτά έχει τον λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως υπόθηκε και ακούστηκε, εκφράζω και εγώ ανησυχία για αυτά που συμβαίνουν στη Συρία. Συνεχίζονται συγκρούσει με αυξανούμενη απώλεια ανθρωπίνων ζώων. Κανένα από τα δύο μέρη δεν μπορεί να επικρατήσει στατιωτικό και η μόνη λύση μπορεί να είναι μόνο η πολιτική λύση που μεταξύ αντιπολίτευση κυβέρνηση θα πρέπει η, η Ευρώπη να κινηθεί προ αυτή την κατεύθυνση. Δεν θέλουμε να κρατήσει ο ο ακραίο και να ικανοποιηθεί η χώρα. Ε, όταν διαλυθούν διάφορες συνιστώσεις εθνοτικές και θρησκευτικέ. Χρειάζεται τοποθέτηση της Ευρώπης σωστή και όπως ήδη άκουσα ήδη γίνεται κάτι τέτοιο, γίνεται επεξεργασία αυτών και ελπίζω να υπάρξουν τα καλύτερα αποτελέσματα για να δικαιωθούν αυτοί οι νεκροί ε, και να σταματήσουν και οι δολοφονίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Απομακρυνόμαστε τώρα από τη λίστα και θα μιλήσει ο κύριος Μπρόκ. Όχι κύριε Χάουιτ, ο κύριος Μπροκ και μετά εσείς. Ε, εμένα να συγχωρείτε λέει ο πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε που μου δώσετε το λόγο γιατί πρέπει έπρεπε να λείψω. Θέλω να κάνω κάποιες ε, παρατηρήσεις. Θεωρώ πως η δουλειά των ε, Υπουργών ε, Εξωτερικών έχει μεγάλη σημασία και η προτομασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αλλά αποδεικνύεται πως η διάσκεψη των φίλων της ε, Συρίας έδειξε σε τι βαθμό είναι κατακαιρματισμένη η αντιπολίτευση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν χρειάζεται να κρίνουμε τον Ασάντο ότι πρέπει να φύγει είναι δεδομένο. Και βεβαίω πράγματι είναι απαράδεκτα αυτά τα οποία γίνονται. Αλλά το αποφασιστικό είναι πως η αντιπολίτευση δεν είναι σε θέση να ενωθεί η δημοκρατική αντιπολίτευση και να έχουν και κάποιο ρόλο οι μειονότητες και φοβούνται οι μειονότητες πως θα υπάρξει μια Ισλαμιστική κυβέρνηση και θα είναι τα πράγματα χειρότερα από ό,τι τώρα για αυτούς και αυτό είναι βασικό πρόβλημα και βλέπουμε πως είναι ένα θέμα το πώς θα κρίνουμε τη χρηματοδότηση από το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία που πάει στα χέρια Σαλαφιστών και Ισλαμιστών. Και αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα. Να πω επίσης πως ε, εκτιμώ την δουλειά των Τούρκων. Η τουρκική κυβέρνηση έχει υπομειστεί μεγάλο βάρος. Φύγεται άμεσα. Η δε κατάρριψη του αεροπλάνου είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να δεχτούμε. Και ο εταίρος Τουρκία σε αυτό το θέμα ως μέλος του ΝΑΤΟ έχει την αλληλεγγύη μας. Αλλά θα ήθελα να επαναλάβω και γνωρίζω ε, πως ο, η είπατε εκπρόσωπος και ο κύριος πρόεδρος του Συμβουλίου θεωρούν πως ε, ο ΑΣΑΔ πρέπει να τελειώσει αλλά ταυτόχρονα πρέπει να βρεθεί μια λύση η οποία δεν θα οδηγήσει σε χειρότερη κατάσταση στην περιοχή και πρέπει να παρακολουθήσουμε μεγάλη προσοχή το ζήτημα αλλά αυτό θα γίνει μόνο αν είναι ενωμένη η δυτική κοινότητα από κοινού με τον αραβικό σύνδεσμο και την Τουρκία. Δεν πρέπει να βγάλουν την ουρά τους απ' έξω οι Άραβες για τις ευθύνες τους για μια ειρηνική ε, λύση με σεβασμό στις μειονότητες. Ευχαριστώ κύριε Μπρόκ. Ακολουθεί ο κύριος Χάουιτ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο Προεδρεύων στη δήλωσή του είπε ότι αυτοί που είναι υπεύθυνοι για τα εγκλήματα θα πρέπει να λογοδοτήσουν. Σας ρωτώ γιατί εσείς και οι συνάδελφοί Υπουργοί Εξωτερικών διέγραψαν την αναφορά για την υποστήριξη την αναφορά στο Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο για τα εγκλήματα που διαπράχθησαν κατά τη ανθρωπότητα ε, που διαπράχθησαν στι Συρίε από το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών. Και γιατί δεν υπευλήθη το κείμενο στον από τη Συρία στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Γενέβη του ΟΗΕ αυτή την εβδομάδα, διότι στην πραγματικότητα δεν υποστηρίζεται με τέτοια αναφορά, τέτοια μνήμα παρά την επανελειμμένη εκκλήση του είπα του εκπρόσωπου του ΟΗΕ αυτό να γίνει. Όπω πολλοί συνάδελφοι σε αυτή τη συζήτηση διαβάσαμε ε, αυτά που ε, είπαν οι υπεύθυνοι για τα δικαιώματα, τα βασανιστήρια που έκαναν συριακές αρχές, ε, χρησιμοποίησαν οξέα από μπαταρίες, σεξουαλικές επιθέσεις, ξυλοδαρμούς, τράβηγμα από τα νύχια, ψευδοεκτελέσεις και το είπε, είπε κάποιος ότι 8 μέρες τον είχαν κρεμάσει από τους καρπούς, δεν μπορούσε να κοιμηθεί, τον αφήνα να κοιμηθεί και είπε ότι σταμάτησε να δουλεύει το μυαλό μου ε, φανταζόμουν πράγματα, ήταν φρικτή η πόνη, ούρλιαζα, έπρεπε να πάω στο νοσοκομείο, αλλά οι φρουροί απλώ γέλαγαν και με κορόιδευαν. Γιατί δεν υποστηρίζετε μία αναφορά στο Εθνικό Δικαστήριο και σήμερα θα δεσμεύσετε την Ευρωπαϊκή Ένωση για κάτι τέτοιο. Ο κύριο Σαλαβράκο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι εξελίξει στη Συρία χαρακτηρίζονται από ένταση τη βία και κλιμάκωση των επιθέσεων τη κυβέρνησης Σάσαντ με βομβαρδισμούς στην πόλη Χόμς και Ντούμα πολλές ανθρώπινες ζωές πάνω από τέσσερις χιλιάδες μέσα στους τελευταίους οκτώ μήνες έχουν χαθεί ενώ ήρθαν παράλληλα στην επιφάνεια φαντάσματα πολιτικών και θρησκευτικών αντιθέσεων και εθνοτικών αντιπαλωτήτων. την ίδια ώρα το κλίμα στα σύνορα με την τουρκία εντείνεται και ανα πάσα στιγμή υπάρχει κίνδυνο στρατιωτικού επεισοδίου ηθελημένου ή αθέλητου. όποιος έχει διαβάσει το βιβλίο στρατηγικό βάθο του νταβούτογλου αντιλαμβάνεται γιατί η τουρκία προσφέρει στήριξη στους σύριους αντικαθεστωτικούς και το έδαφος της αποτελεί έδρα πολλών αντικαθεστωτικών ομάδων και δι' ασυντόνιστων όπως επεσήμανε και ο κύριος υπουργός στην πρωτολογία του. οι χριστιανοί στην περιοχή αισθάνονται ανασφαλείς στο μέτωπο της διεθνούς διπλωματίας η διαμάχη ρωσίας δύσης παραμένει και η μόσχα αρνείται να παραστεί στη σύνοδο των φίλων της συρίας την επόμενη παρασκευή. μια παγκόσμια κρίση ελοχεύει και παρακαλώ πρέπει να την προσέξουμε. ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Σαλαβράκο. Ο κύριος Αγκουράκης για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ζητώ συγγνώμη ε, καταγγέλνουμε τις αποφάσεις του ευρωπαϊκού συμβουλίου της 29 του ιουνίου για τη συρία και το ιράν γιατί σηματοδοτούν κλιμάκωση της υπεραλιστικής επέμβασης της ε, ε, ευρωπαϊκής ένωσης των ηπα και του νατο στην περιοχή στο έδαφος σκληρών ανταγωνισμών με τις καπιταλιστικές δυνάμεις της ρωσίας της κίνας και της ινδίας. δυναμώνει απειλές των ηπα και του νατο αλλά και της τουρκίας του κατάρ της σαουδικής αραβίας του ισραήλ στην περιοχή αυτή τη στιγμή αεροπλανοφόρα των ηπα συγκεντρώνονται στην περιοχή και αυξάνεται η κινητικότητα στη βάση της Σούδα στην ελλάδα. εξετάζεται η επιβολή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων με πρόσχημα την ευθύνη την προστασία των αμάχων που χρησιμοποιήθηκε και σε άλλες συμβιβαστικές επεμβάσεις. οι ηνωμένε πολιτείε το νατο και η ευρωπαϊκή ένωση κράτη της περιοχής επεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις της συρίας παραπληροφορούν εκμεταλλεύονται τη σύγκρουση να δικαιολογήσουν ένα νέο πόλεμο. οι εξελίξεις στη συρία συμπληρώνουν την κατοχή στο ιράκ στο αφγανιστάν και στη λιβύη καταγγέλνουμε επίσης τις αποφάσεις του νάτο το οποίο με πρόσχημα της δίθεν ε, ατλαντικής αλληλεγγύης στην τουρκία πρωτοστατεί στην υπερελιστική αρμάδα κατά της συρίας για στρατηγικό πλήγμα και κατά του ιράν. εντείνονται οι κυρώσεις και η ευρωπαϊκή ένωση απειλεί με ανοιχτή στρατιωτική επέμβαση αν δεν περάσουν τα υπερελιστικά σχέδια για ανατροπή της συριακής κυβέρνησης από τις 1 Ιουλίου, όπως γνωρίζουμε, εφαρμόζονται αποφάσεις για επιβολή εμπάργκο στο πετρέλαιο από το Ιράν με ε, ολέθριες συνέπειες. Οι εξελίξεις στη Συρία αφορούν τον λαό της Συρίας. Είναι ανάγκη οι λαοί να αντισταθούν στις επεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και να ανατρέψουν τα υπεραλιστικά σχέδια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε κύριε Αγκουράκη. Ο κύριος Αλχαντράουι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρέπει να τελειώσουν οι ακρότητες στην ε, Συρία. Αλλά από ό,τι φαίνεται ε, η διεθνής κοινότητα μόνο κοιτάει. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε τη συνάντηση της ε, Γενέβης ως ε, επιτυχία. Και από ό,τι φαίνεται η μόνη πραγματική λύση είναι διαπραγματεύσει μεταξύ του καθεστώτος και της αντιπολίτευσης. Αλλιώς η εναλλακτική είναι ένα εμφύλιος πόλεμος, αλλά βεβαίω η κατάσταση είναι ανησυχητική. Θα πρέπει λοιπόν η διεθνή κοινότητα να φέρει κυβέρνηση και αντιπολίτευση γύρω από το ίδιο τραπέζι. Συμφωνώ με τον κύριο Μπρόκ πως ε, ουσιαστική ε, προϋπόθεση για την επιτυχία και για την αντιπολίτευση είναι να, φιλήσει, να μιλήσει με μία φωνή. Να έχει ένα όραμα για το μέλλον της Συρίας και βεβαίως να καθησυχάσει αυτούς οι οποίοι αμφιβάλλουν για ε, την στήριξη του καθεστώτος. Οπότε θα ήθελα να ζητήσω να παραμείνει η πίεση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ελ Χαντραουή. κυρία Ερτσούκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, η κατάσταση στη Συρία όλο και επιδεινώνεται παρά τις προσπάθειες που γίνονται σε διεθνές επίπεδο για την εξέβρεση λύσεως μέσω διαπραγματεύσεων και κινδυνεύει η κατάσταση να επιδεινωθεί μετά την κατάρριψη του ε, τουρκικού αεροσκάφους. Πεθαίνουν καθημερινά αθώοι σαν αποτέλεσμα φρικτών σφαγών που ε, είναι κατά του λαού της Συρίας που θέλει να ζήσει δημοκρατικά και η μεταφορά όπλων εκεί στη χώρα δείχνει ότι γίνεται πιο επικίνδυνη η κατάσταση. Να μην μιλήσουμε για την κατάσταση των χριστιανών. Και η θέση της Ρωσίας και της Κίνας δυστυχώς είναι κατηγορηματική. Δεν δέχονται τίποτα που να αφορά την αλλαγή του πολιτικού καθεστώτος και συμφωνώ με τα εδώ υποθέντα, δηλαδή ότι είμαστε υπεύθυνοι για την προστασία των θυμάτων. Εκτιμώ τη θέση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που δρά συνεκτικά για την εξέβρεση ειρηνικής λύσης. Θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες ούτω ώστε να διαπραγματευτούμε την λύση της κρίσης αυτής μεταξύ κυβερνήσεων και πολίτευση και η ειρηνική λύση. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Κρετσού. Ο κύριος Ρωμένο Λόπες για ένα λεπτό. Κυρία Ρομέρα Λόπε, συγγνώμη, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένα από τα στοιχεία τα βασικά του σχεδίου του Κόφι Ανάν είναι η αποχώρηση των ε, στρατιωτικών δυνάμεων στους ε, στρατώνες τους. Αυτή είναι μια κοινή γραμμή που ακολουθούν όλες οι χώρες για να αποφύγουν την έκρηξη ενός εμφυλίου πολέμου στην Συρία. Είναι γεγονός πρέπει να εργαστούμε ώστε να υπάρξει συνεκτικότητα και συνοχή Τη αντιπολίτευση στη Συρία. Είχαμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρουσία εκπροσώπων από το Συριακό Εθνικό Συμβούλιο και προσπαθήσαμε να το επιτύχουμε αυτό, αλλά είναι απαραίτητη και η πίεση τη Ευρωπαϊκής Ένωσης για το εμπάργο όπλων και την πραγματική εφαρμογή αυτού του μέτρου. Τι συνέχεια δίνει στα θέματα αυτά το Συμβούλιο. Τι πληροφορίες έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την εφαρμογή αυτού του εμπάργου, τι ε, έχουν συσσωρεύσει κυβερνητικέ δυνάμεις. Μπορεί πράγματι να συνεχίσει η Ρωσία να εφοδιάσει με όπλα τη Συριακή κυβέρνηση, γιατί είναι δύσκολη η διαπραγμάτευση με τη Ρωσία, αλλά είναι απαραίτητο για το θέμα αυτό να έχουμε την βεβαιότητα ότι δεν θα <clears throat> πάει ο στρατό στους στρατώνε του και δεν θα έχει και περαιτέρω εξοπλισμό. Ευχαριστούμε κυρία Ροπέρο Λόπες. Ερχόμαστε στην διαδικασία Catch the Eye. Ο κύριος Σόνικ. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε. Όλοι έχουμε νιώσει συντριβή βλέποντας αυτά που συμβαίνουν στη Συρία. Νομίζω ότι το κλειδί για την αποφυγή περαιτέρω αιματοχυσίας είναι βέβαια δράση που θα αναλάβει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Γι' αυτό θα πρέπει να υποθεί ξεκάθαρα ότι η παρούσα, το παρόν αδιέξοδο είναι αποτέλεσμα κινήσεων που μπλοκάρουν τις προσπάθειες και την, μπλοκάρουν τις προσπάθειες η, Ρωσία και η Κίνα. Και θα πρέπει να σκηθούν πιέσεις προς τα εκεί από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα πρέπει να εθελοτυφλούμε ε, όσον αφορά τα όσα κάνει η Μόσχα. Ε, η Μόσχα θα μπορούσε αμέσως να σταματήσει την αιματοχυσία. Μέχρι τώρα οι προσπάθειες που κάναμε δεν έδωσαν αποτελέσματα ο Ρώσος Υπουργό Εξωτερικών κάνει ότι, ότι αναλαμβάνει κάποια δράση και μόνο αυτό κάνει. Μόνο η διεθνής υπεροή και πίεση επί της Μόσχας να αναλάβει δράση επί τόπου θα είναι αποτελεσματική λύση και διέξοδος από την κρίση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Σόνικ. Ακόμα και αν μπορούμε να, έχουμε ο καθένας μας τις απόψεις μας για τη δυνατότητα διευθέτησης του προβλήματος με διπλωματικό ή πολιτικό τρόπο θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα προφανώς ούτως ώστε η συμφωνία της Γενέβης να εφαρμοστεί ελπίζω ταυτόχρονα θα πρέπει να κανουμε τα παντα προφανως Συρία, ωστε η συμφωνια της γενεβης να εφαρμοστει ελπιζω ταυτοχρονα θα πρεπει να υποστηριξουμε τη Συρια... την αντιπολίτευση της Συρίας ε, να υποστηρίξουμε την ενότητά τη, να αντιμετωπίσουμε την ανθρωπιστική κρίση, κάτι που κάνετε, να ρίξουμε φω, άπλετο φω στα όσα συμβαίνουν στη Συρία, κάτι που ζήτησε είπα ω εκπρόσωπο του ΟΗΕ και έχει δίκιο και μπροστά στι φοβερέ διαπιστώσει των μη κυβερνητικών οργανώσεων, και είδατε όλη αυτή την έκθεση, το αρχιπέλαγο των βασανιστήριων ήταν ο τίτλο, θα πρέπει να μα οδηγήσει να σκεφτούμε, να, δούμε, να αλλάξουμε πώ λειτουργεί το Συμβούλιο Ασφαλεία στο ΙΕ. Από την πλευρά μου, όταν πρόκειται για καταδίκη όσον αφορά τα εγκλήματα τη ανθρωπότητα, δεν θα πρέπει να υπάρχει το δικαίωμα αρνηση ούτε μπλοκάρισμα. Θα πρέπει να γίνεται κάτι τέτοιο από την πρώτη στιγμή. Ευχαριστώ. κυρία Κύριε Στάνο, για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, λένε τώρα οι επικεφαλής αντιπολίτευσης Συρίας πως 15.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη σύγκρουση που διαρκεί 1,5 χρόνο και οι λιποτάκτες από τις δυνάμεις του Ασάντ επιβεβαιώνουν αυτά τα νούμερα. Το Εθνικό Συριακό Συμβούλιο με τους Ισλαμιστές αλλά και άλλες κοσμικές αντιπολιτευτικές ομάδες πρέπει να ενωθούν τώρα κατά του μπαθικού καθεστώτος του Ασάντ ενώ πλέον έχουμε χαρακτηριστικά εμφυλίου πολέμου στην σύγκρουση. Η ύπατη εκπρόσωπος πρέπει να στηρίξει τη Συμφωνία της Γενέβης για να έχουμε μια μεταβατική κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας πλην ε, Ασάντ για να ανοίξει ο δρόμος για δημοκρατικέ εκλογέ. Το σχέδιο Ανάν ίσω αποδειχτεί επιτυχία. Δράτω με τις ευκαιρία να ευχαριστήσω και την Τουρκία για τη βοήθειά τη με τους πρόσφυγε και στέλνω τα συλληπιτήριά μου στους ε, οικογένειε των πιλότων που καταρρίφθηκε, του αεροπλάνου που καταρρίφθηκε από τις, ε, το Συριακό Σύστημα Εράμινας. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να τερματιστεί αυτό το φρικτό καθεστώ στην Δαμασκό. Επιτρέπετε κύριε Τανόκ μια ερώτηση από τον κύριο Χάουιτ. Κύριε Χάουιτ, Ευχαριστώ. Ξέρω πως ο αγαπητός συνάδελφος έκανε την δήλωσή του με να, τον ρωτήσω γιατί η δική μας η κυβέρνηση υπό την ηγεσία του κόμματός του δεν συντάχθηκε με όλες οι υπόλοιπες χώρες για να γίνει ακριβώς αυτή η αναφορά στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο καθώς θα μπορούσε να πει κανείς πως καθυστέρηση δημιουργούσε τις πιθανότητες μιας λύσης, αλλά δεν έγινε αυτό, ανταυτού είχαμε περισσότερες παραβίασεις των ορισμένων δικαιωμάτων. Γιατί δεν έκανε αυτή την έκκληση η Μεγάλη Βρετανία. Απάντηση. Ο κύριο Χάουτ ξέρει πολύ καλά πω δεν εκπροσωπώ τη Βρετανική κυβέρνηση. Είναι μια συμμαχική κυβέρνηση. Δεν είμαι εγώ υπόλογο για το τι κάνει το Υπουργείο Εξωτερικών ή ο Πρωθυπουργό. Το μόνο μπορώ να πω είναι πω θα ήθελα να δικαστεί ο κύριο Ασάντα από το Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο, αλλά ίσω θα μπορούσε να είναι θετικό να δώσουμε την ε, ευκαιρία στον ε, κύριο Ασάντ να φύγει από την εξουσία γιατί αν ε, θεωρεί πως μπορεί να δικαστεί ίσως προκαλέσει μεγαλύτερη αιματοχυσία. Θα μπορούσαμε λοιπόν να του δώσουμε μια διέξοδο να φύγει από την Δαμασκό και να πάει στην εξορία. Υποθέτω. Ευχαριστώ κύριε Σπέλτερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. ήθελα να ε, υποβάλω κάποιες σκέψεις στους εκπροσώπους του Συμβουλίου. Δεδομένης δραματικής κατάστασης ε, στην Συρία, βεβαίω θα πρέπει να υποστηρίξουμε ε, μια λύση η οποία θα είναι διαθρησκευτική, διαεθνοτική και ελπίζω βεβαίως να τα κάνει αυτά η προσωπία μας στην ε, Δαμασκό πρώτον και δεύτερον. Μιλήσαμε για την ε, παρακολούθηση της κατάστασης των χριστιανών. Αν δείτε το τι συμβαίνει στην Χόμς υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ενισχύα και υπάρχουν και κάποιοι Σουνίτες ε, εκεί πέρα και μιλάμε για απαγωγές ε, και ζητάνε μετά παράλογα λίτρα, δολοφονούνται ψυχρό ιερείς. Είναι λοιπόν πραγματικά δραματική η κατάσταση και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δει το τι γίνεται εντός της Συρίας και να μην ασχολείται μόνο με την αντιπολίτευση που βρίσκεται εκτός της χώρας. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Όμπερμαϊρ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε ακούμε τις ιστορίες φρίκης για φόνους, για, για βασανιστήρια κτλ. Η ανθρωπιστική βοήθεια, όσο σημαντική και να είναι και όσο να συμβάλλει, δεν μπορεί ποτέ να επιλύσει το ίδιο το πρόβλημα. Όσο υπάρχει, αυτό το, όσο υπάρχει αυτή η κατάσταση, έχουμε να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο την κυβέρνηση του Βασίρα Αλασάτα, αλλά και τι Ισλαμιστικές ομάδε, οι οποίε υποστηρίζονται από την Σαουδική Αραβία και είναι τμήμα μια κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση. Είδαμε ότι συναντήθηκε η αντιπολίτευση με την αδελφότητα των μουσουλμάνων στην Αίγυπτο και φοβόμαστε ότι υπάρχει πραγματικά ένα πρόβλημα για την χριστιανική μειονότητα στη Συρία, που είναι της τάξης του 15%. Δεν μπορούμε λοιπόν να υπάρξει καμία μετάβαση χωρίς μια πραγματική συμμετοχή στις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας από τη Ρωσία. Πρέπει λοιπόν να επιζητήσουμε την, ε, την λύση για να μην δημιουργηθεί μια κατάσταση χάους όπως το Ιράκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ομπερμάιερ. <clears throat> Κλείνουμε την κυρία Όουλαντ ως τελευταία ομιλήτρια στη διαδικασία Κατσδία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να χαιρετήσω Καλωσορίζω λοιπόν το αποτέλεσμα τη συνεδριάσεω τη ομάδα δράση για τη Συρία και την υποστήριξη του ειρηνευτικού σχεδίου του Κόφια Ανάν. Ο καταστροφικό εμφύλιο πόλεμο που θα επηρέαζε όλη την περιοχή δεν είναι εναλλακτική λύση όσον αφορά τη διπλωματική προσέγγιση. Ελπίζω ότι όλα τα μέλη τη ομάδα δράση ότι θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να εφαρμόσουν το τελικό ανακοινωθέν. Τα εμπόλεμα μέρη πρέπει να σταματήσουν κάθε βιοπραγία, ώστε διαπραγματεύσει για το μέλλον του λαού τη Συρία να μπορέσουν να ξεκινήσουν. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα πρέπει να συνεννοηθούν μεταξύ τους και να έχουν αίσθημα ευθύνης όσον αφορά τον Συριακό λαό, τόσο ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία τη διαμόρφωση μια μεταβατική κυβέρνηση, σχηματισμού μεταβατική κυβέρνηση. Οπότε θα αρνείω την είπατε εκπρόσωπο να επιμείνει, ούτω ώστε όλα τα κινήματα αντιπολίτευση τη Συρία που αντιμετωπίζουν εθνοτικέ, ε, ε, διαφορετικέ συνιστώσει σκεφτικέ και εθνοτικέ, να μπουν στι διαπραγματεύσει, ούτω ώστε να γίνει μια βιώσιμη μετάβαση από αυτό το καθεστώ σε ένα άλλο. Ευχαριστώ. ευχαριστώ για να ολοκληρώσει την συζήτηση ακόμη μια φορά ο κύριος Μαυρογιάννης έχει το λόγο Thank Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε Πολλοί αγορητές αναφέρθηκαν στο σεβασμό των μειονοτήτων και κυρίως των θρησκευτικών και πιο ιδιαίτερα αναφέρθηκαν στις χριστιανικές μειονότητες και σας διαβεβαιώ ότι υποστηρίζουμε όλες τις ομάδες που εργάζονται για την ειρήνη και παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς ε, την κατάσταση που επικρατεί για κάθε τέτοια ομάδα και από τις πολλές κοινότητες που υπάρχουν στη Συρία που σημαίνει χριστιανικές κοινότητες επίσης και πάνω απ' όλα. Παρατηρούμε τι γίνεται λοιπόν. αναφισβήτητα τα ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται στην ε, Συρία, όμως αληθεύει ότι η αναφορά στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο γνωρίζουμε όλοι πόσο είναι ένα επίτευγμα διεθνού κοινότητα στο Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο και πόσο το εκτιμούμε και πόσο πολύ πιστεύουμε στη λογοδοσία. Όμως αληθεύει ότι μηνύα του Διεθνού Ποινικού Δικαστηρίου και στη Γενέβη αλλά και στη Νέα Υόρκη όπου συζητείται το νέο ψήφισμα η μηνύα αυτή λέγω ήταν στο επίκεντρο συζητήσεως τα κράτη-μέλη συζητούσαν αν ήταν η σωστή στιγμή και αν ήταν σκόπιμο να υπάρξει τέτοια μνήμα και τέτοια αναφορά. Τώρα που όλοι προσπαθούμε να δώσουμε νέα όθηση στην αποστολή του Κόφι Και θέλουμε και η Ρωσία και η Κίνα να υποστηρίξουν τη νέα ομάδα δράσης και το νέο δικό χάρτη. Συμφωνήσαμε όλοι τώρα να αποφύγουμε τώρα, αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη φάση, τώρα, σε αυτό το στάδιο, το υπογραμμίζω, ή αδίποτε επίμαχα ζητήματα. Όμως σίγουρα θα πρέπει να επιστρέψουμε στο θέμα αυτό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Θα ήθελα να πω επίσης ότι ακούσαμε με μεγάλο ενδιαφέρον αυτή τη σημαντικότητα της συζήτηση μαζί με τον καλό μου φίλο, τον Γενικό Γραμματέα τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία εξωτερική Δράσης, τον Πιέρ Βημών, και θα ενημερώσουμε δεόντως την ύπατη εκπρόσωπο και αντιπρόεδρο ε, Άστον. Για αυτά που υποθήκαν, προσβλέπουμε σε περαιτέρω συζητήσει όσον αφορά την κατάσταση στη Συρία τι επόμενε εβδομάδε και του επόμενου μήνε. Όσο συνεχίζεται αυτή η μεταβατική διαδικασία, θα σα ενημερώνουμε δεόντω για τι δράσει τη Ευρωπαϊκή Ενώση σχετικά με το θέμα. Με την υποστήριξή σας ελπίζουμε ότι οι διεθνείς δράσεις θα αποδώσουν καρπούς και θα σταματήσει η βία η καταστολή στη Συρία και θα επιτραπεί μια ειρηνική και δημοκρατική μετάβαση. Σας ευχαριστώ αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου για την υποστήριξή σας, για τις ερωτήσεις σας και για τις ανησυχίες που εκφράσατε. Όλα αυτά συμβάλλουν στον καθορισμό της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σε αντίδραση στην κρίση στη Συρία. Σας καλούμε να παραμείνετε αφοσιωμένοι σε αυτό το σκοπό, ώστε όλοι οι πόροι μας, όλες οι ιδέες μας να χρησιμοποιηθούν στο μέγιστο βαθμό. Θα ήθελα τώρα, επειδή μου ζητήθηκε, να απαντήσω υπό την εθνική μου ιδιότητα σε ερώτημα, σαν εκπρόσωπος της κυβερνήσεως της Κύπρου, να σας απαντήσω για το θέμα των κυρώσεων και το συγκεκριμένο ζήτημα του πλοίου ε, που ελιμενίστηκε που μετέφερε τα όπλα. Λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι η Κύπρος σέβεται και εφαρμόζει πλήρως το εμπάργκο των όπλων που ισχύει ε, τη Συρία και για άλλες χώρες που έχουν υποστεί κυρώσεις και τονίζει περαιτέρω τη σημασία συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για αποτελεσματικότερη εφαρμογή ε, του εμπάργου όπλων και αποδεικνύει ότι είναι έτοιμη να ξεκινήσει σχετική συζήτηση στα ενδεδειγμένα βήματα για να καθοριστούν οι βέλτιστες δυνατές πρακτικές. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση με το σκάφος Chariot, θα ήθελα να υπογραμμίσω τα εξής. Οι λιμενικές αρχές της Κύπρου έλαβαν διαβεβαιώσεις από τον πλοίαρχο του εν λόγω πλοίου και από την πλειοκτήτρια εταιρεία ότι τελικός προορισμός του φορτίου ήταν το Ισκεντερούν στην Τουρκία και όχι Συρία. Όλοι γνωρίζουμε μετά τι συνέβη. Όμως μετά αυτό το γεγονός και η μερική αστυνομία του Ισκύπρου και οι τελωνιακές αρχές εξέδωσαν νέες εγκυκλίους υπενθυμίζοντας στο προσωπικό και όλες τις πλειοκτήτες εταιρείε την ύπαρξη των περιοριστικών μέτρων και των κυρώσεων κατά τρίτων χωρών και πιο συγκεκριμένα κατά της Συρίας και κατά του Ιράν. Και προειδοποιούσαν ότι θα υπάρχουν νομικές συνέπειες σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Η λιμενική αρχή της Κύπρου ήδη έδωσε οδηγίες στους ε, δικηγόρους της να ξεκινήσουν ποινικέ διαδικασίες κατά της πλειοκτήτριας εταιρεία και του πλειάρχου του σκάφους αυτού. Η Δημοκρατία της Κύπρου τονίζει ότι είναι πλήρω δεσμευμένη στην εφαρμογή των μέτρων τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και των κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλεία κατά τρίτων χωρών. Επαγρυπνούμε. Θέλουμε να εφαρμόσουμε πλήρω το εμπάργκο όπλων τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω κατά τη Συρία και κατά άλλων απολυταρχικών καθεστώτων. Και γι' αυτό προσβλέπουμε σε επικοδομητική συνεργασία με τους εταίρους της Ευρωπαϊκής με ε, κοινοποίηση γνώσεων, πληροφοριών και είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε στη συλλογική διεθνή προσπάθεια για να, μη, να μειωθεί η διάδοση των όπλων, νέων τεχνολογιών και να θέλουμε να προωθούμε την ειρήνη, σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό γίνεται έτσι σημαντικότερο λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωγραφική θέση της Κύπρου είναι πολύ κοντά στην περιοχή αυτή ε, των αναταραχών στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Και είμαστε και κόμβος ε, όσον αφορά την αυσιπλοεία. Άρα εκεί απαιτείται ιδιαίτερη επαγρύπνηση όσον αφορά τις προσπάθειες να εφαρμόζουμε τους περιοριστικούς όρους, τα μέτρα, τα περιοριστικά ε, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Μαυρογιάννη. Έχει κλείσει η συζήτηση λοιπόν για το θέμα αυτό κάποιες ανακοινώσεις από το ΕΛΚ και το ΙΕΦΤΕ. Έχω